Uh, uh, um, Καλημέρα σας κυρίε και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινούμε την δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους επισκέπτες μας, γιατί έχουμε μια ομάδα επισκεπτών από την τουρκική αρχή ανταγωνισμού, που είναι εδώ παρόντες ως ε, τμήμα μιας ε, διαδικασίας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης και θέλουν να μάθουν περισσότερα για το δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήλθατε λοιπόν ως Κελτινής και δεν θα αντιμετωπίσουμε μεν τα θέματα του δικαίου ανταγωνισμού, αλλά θα έχουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην έκθεση του κυρίου Μπουζόιλ που αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 θα έχουμε μια ειδική παρουσίαση μελετών για τον αντίκτυπο της ε, διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν ως τμήμα της εργασίας του κ. Ζουβέν για τον αντίκτυπο, που κάνει ο κ. Ζουβέν για τον αντίκτυπο της διαφήμισης στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Από τις 11 θα ξεκινήσει αυτό. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο στον κ. Μπουζόιλ να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε μια συνάντηση στο συντονιστό για μια μισή ώρα σήμερα το πρωί για να συζητήσουμε μια σειρά από στρατηγικού χαρακτήρα θέματα τα οποία θα σταλούν στα μέλη της Επιτροπή μας. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα μετά από σήμερα βέβαια το πρωί και το απόγευμα θα είναι την 5η 2 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί και εκεί θα εγκρίνουμε την έκθεση της κυρίας Ρίλε για τον προϋπολογισμό και επίσης του κυρίου Κορέα Δεκάμπους. Αυτά λοιπόν για την ημερήσια διάταξη της Δευτέρα Σεπτεμβρίου και θα υπάρξει και μια ειδική και κλεισμένη των θυνών συνάντηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Περνάω λοιπόν τώρα στην γνωμοδότηση της Επιτροπής μας σε σχέση με την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση του κοινοτικού δικαίου, 26η ετήσια έκθεση. Ο κύριος Μπουζόη είναι ο εισηγητής και μετά θα ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών και των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε λοιπόν με τον εισηγητή τον κύριο Μπουζόη και η κυρία Ράπτη επίσης είναι παρούσα, η κυρία Ρούλε. Δεν βλέπω άλλους ε, σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες. Ίσως θα έρθουν στη συνέχεια. Ίσως και το ΕΛΚ θα στείλει κάποιον για να κάνει κάποια σχόλια. να έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η 26η ετήσια έκθεση για, την, για τον έλεγχο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από την μη έγκαιρη και μη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Το πρόβλημα δεν είναι η, γνώση, αν θέλετε, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αυτή καθεαυτή, αλλά ε, το κατά πόσον οι καταναλωτές και οι πολίτες μας μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια τα οποία προσφέρει, θα μπορούσε να τους προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Μάριο Μόντι προσπαθεί να ε, βελτιώσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί καλύτερα, ε, πιο σωστά η εσωτερική αγορά. Έχω προτείνει κάποιες ε, προτάσεις στην έκθεσή μου που εμπνέονται από τις προτάσεις ε, του Μάριο Μόντι. Οι πολλές ιδέες προτέλθουν από τις τροπολογίες, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτες οι τροπολογίες και από τους άλλους συναδέλφους, αλλά και από τους σκιώδες εισηγητές. Ε, θα ήθελα να επίσης να τονίσω και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Έχουμε αυξήσει τις ε, διαδικασίες ε, παράβασης λόγω της μη εφαρμογής, έγκαιρης εφαρμογής της και μετάθεσης της κοινοτικής νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη έχουν να, βέβαια να μεταθέσουν στην εθνική νομοθεσία λιγότερε οδηγίε από το 2007. Έχουμε προβλήματα όμω στον τομέα των υπηρεσιών. Το συζητήσαμε, ε, έχουμε συζητήσει ήδη και για την εφαρμογή τη οδηγία ε, για τι υπηρεσίε, για τα επαγγελματικά προσόντα. Επίση ε, έχουμε το πρόβλημα των δημοσίων κρατικών προμηθειών και έχουμε επίση και νομοθεσία που ε, υιοθετείται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μετατίθεται και δεν εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως ε, είναι και μια πιο θετική ε, στάση από πλευράς των κρατών μελών. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι περίπλοκο θέμα. Διότι αν δεν μεταθέσουμε τις οδηγίες έγκαιρα, τότε εμποδίζουμε ε, τους πολίτες να απολαύσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για κάτι άλλο. Δεν κατηγορώ μόνο τα κράτη-μέλη, διότι στο κάτω-κάτω δεν είναι και τα μόνα υπεύθυνα. Γι' αυτό ακριβώς όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε τις δεσμεύσει μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τα κοινοτικά όργανα θα πρέπει να ε, εναρμονίσουν και να συντονίσουν τις στάσεις τους έτσι ώστε να προωθηθεί και η καλύτερη ε, εφαρμογή και μεταφορά της νομοθεσίας θα πρέπει επίσης να, συντο... να ενδυναμωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Να εξηγούμε πλήρως τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Το φόρουμ για την ενιαία αγορά το οποίο θα οργανώσουμε το φθινόπωρο και ελπίζω ότι θα είναι ένα ετήσιο μεγάλο συμβάν της μας σε συνεργασία με την Κομισιό και το Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελέσει και ε, ένα έναυσμα για να βελτιωθεί η κατάσταση και να συζητήσουμε την, ε, και τα θέματα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίση, θα ήθελα να τονίσω την σημασία της ε, ε, των υπηρεσιών ε, εξυπηρέτηση αν θέλετε της εσωτερικής αγοράς. Ε, θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα το Europortal και άλλα project αντίστοιχα και παρόμοια, διότι είναι ζωτική σημασία για τους καταναλωτές και τους πολίτες μας να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά και να έχουν τα εργαλεία τα, στη διάθεσή τους όπου θα τους είναι αναγκαία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τις απόψεις για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα η γνωμοδότηση θα, θα ψηφιστεί στις 13 Σεπτεμβρίου, έτσι είναι προγραμματισμένο. και αυτό θα ήθελα να προτείνω σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, να το δούμε, ε, να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες, να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής μας, τη ΣΥΜΚΟ, για την δουλειά που έχει κάνει και Θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Το περιμένω με ανυπομονησία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουζόη. Κύριε Σώση, θέλετε Θέλετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας πριν σας δώσω το λόγο. Η κυρία Ράπτη, η κυρία Ράπτη είσαστε κι εσείς σκιώδης συγητής. Θα, δώσετε το, θα σας δώσω το λόγο τώρα. Η ε, κυρία Οτσακόφσκη, η κυρία Μιούλερ. Δεν ξέρω κανείς άλλος ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Η κυρία Ράπτη τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπουσό για τη δουλειά που έχει κάνει. Ε, έχω παρακολουθήσει τη δουλειά που έχει κάνει όπως όλοι μας άλλωστε και σε προηγούμενες εκθέσεις και πραγματικά η τεκμηρίωσή του βοηθάει πάρα πολύ τη δουλειά μας. Ε, το κείμενο το οποίο μας παρουσίασε είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης. Θέλω να επισημάνω ορισμένα σημεία. Ε, μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής του δικαίου του ευρωπαϊκού. Είναι σημαντικοί όσοι ακόμη δεν έχουν επαρκώς εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός αμοιβαίας αξιολόγησης στην οδηγία για τις υπηρεσίες, ε, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστούν και στη συνέχεια να δούμε εάν και πώς θα πρέπει να επεκτείνουμε την εφαρμογή τους. Ε, επιμένω ιδιαίτερα στο να έχουμε αξιολόγηση ε, όσων μηχανισμών λειτουργούν, γιατί νομίζω ότι αυτό θα κάνει τους μηχανισμούς να λειτουργούν όχι μόνο για να λειτουργούν και να υπάρχουν, αλλά για να είναι προς όφελος ε, των πολιτών. Εξάλλου πιστεύω ότι σκοπός όλων μας είναι η αποτελεσματικότητα και όχι η δημιουργία περισσότερης γραφειοκρατίας και των αγγυλώσεων που προκύπτουν από τη γραφειοκρατία ε, πειραματικοί μηχανισμοί που έχουν ήδη φέρει πρώτα θετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το EU Pilot. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρώ επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνέργειες μεταξύ των εθνικών διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα, και στο τοπικό και στο εθνικό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η θέσπιση ενός πάγιου αιτήματο των πολιτών, ενός πάγιου αιτήματο των καταναλωτών και μιλώ για τον μηχανισμό συλλογικών προσφυγών και συλλογικών αποζημιώσεων που θα πρέπει να τον δούμε ως ένα ε, δημοκρατικό μέτρο που τονώνει την κοινωνική συνοχή και δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά στο πλευρό των πολιτών. Και αυτό γιατί ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους με τη συμπεριφορά τους βλάπτουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ε, θέλω να επισημάνω ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάζει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία επιπαραβάση όπου χρειάζεται. Και ναι μεν εδώ μιλώ εκ μέρους των σοσιαλιστών, αλλά ταυτόχρονα είμαι και Ελληνίδα. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ στον τομέα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Άρα ε, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία ε, το γεγονός ότι τονίζω πως η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάζει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία επί παραβάση όπου χρειάζεται. Τέλος, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί και πρέπει να πιέζει περισσότερο την Επιτροπή τόσο για να παρακολουθεί την εφαρμογή ε, του κοινοτικού δικαίου στις χώρες μέλη, όσο και για την επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Ε, συνάδελφε, δεν θα μιλήσω τώρα για το θέμα των τροπολογιών, που είναι πάρα πολύ αξιόλογες, και έχω μερικά ε, σημεία να επισημάνω, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα ε, να τα πούμε στις 5 η ώρα στην συνεδρίαση των σχεδόν, έτσι όπως ακριβώς είπατε με λεπτομέρειες, ώστε να προετοιμάσουμε το δυνατόν καλύτερα τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ και πάλι για την δουλειά και το πολύ καλό κείμενο βάσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, thank you, Mrs. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ράπτη. Κύριο Τσερκόφσκι. Συγγνώμη που καθυστέρησα κύριε Πρόεδρε, ήμουν στην Συνταγματική επιτροφή που είμαι υποσυντονιστής του ΕΛΚ και είχα μια συνάντηση με τη Βελική Προεδρία εκεί. Συγχαρητήρια καταρχήν για το πολύ καλό έργο το οποίο έχετε κάνει. Γενικά, μπορούμε να εξάρουμε την ε, γνωμοδότηση αυτή, το σχέδιο γνωμοδότηση γιατί είναι συνοπτική και αντιμετωπίζει όλα τα ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, ιδίως από την οπτική γωνία της Επιτροπής μας και είναι σύντομη και περιεκτική αυτή η γνωμοδότηση και εύστοχη και εστιάζει στην, στους εσωτερικούς μηχανισμούς, στον διαθεσμικό διάλογο κτλ. Το μόνο πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχουμε μερικές από τις τροπολογίες είναι ότι κάποιες από αυτές, ιδίως προς το τέλος, μπαίνουν στην ουσία για θέματα παραγωγικά δημόσιων προμηθειών. που προσπαθείτε να συνοψίσετε εκεί την θέση τη Επιτροπής μας για θέματα δημοσίων προμηθειών ή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, που μερικές φορές όμως μπορεί τα σημεία αυτά να είναι επίμαχα μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας σε κάποιες επίσης από τις τροπολογίες σας που είναι θαυμάσιες ουσιαστικά εξετάζεται την ουσία της ε, έκθεσης. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε τόσο πολύ σε βάθος και να ασχοληθούμε με την ουσία της έκθεσης σε τέτοιο βάθος και έκταση. Μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε περισσότερο όταν συναντηθούμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση και οι περισσότερες τροπολογίε κινούνται προ την σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να καταλήξουμε λοιπόν σε μια καλή συμβαστική λύση και επομένως η γνωμή τη Επιτροπής μας για το πώς <clears throat> γίνεται η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Κυρία Ρούλιο, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι μια πολύ καλή έκθεση θέλω να τονίσω αυτά που λέει ιδιαίτερα στο σημείο 3. Το θέμα των πινάκων συσχετισμού. Είχαμε πάντα πολλά προβλήματα γιατί το Συμβούλιο δεν δέχτηκε τη σημασία αυτών των πινάκων. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω ιδιαίτερα το σημείο 3 του εισηγητή. Έχω μια παρατήρηση στο σημείο 5. Είναι <clears throat> θετική αυτή η διαδικασία αλλά θα έχουμε ήδη κάποιες αναφορές από πολίτες που λένε ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική. Όταν πρόκειται λοιπόν για κάποια έστω και μικρή αλλαγή μιας ε, ρήτρα θα πρέπει να μπαίνουμε σε ένα τόσο μεγάλο γραφειοκρατικό επίπεδο. Κάπου θα πρέπει να θέσουμε τα όρια ώστε αυτό να οδηγήσει σε σαφήνεια και για την Κομισιόν και για τις υπηρεσίες σε χαμηλότερο επίπεδο που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε σαφή όρια ώστε να μην οδηγήσουν αυτά σε υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος και να εμποδίσουν να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Το σημείο 8 επίση μου φαίνεται πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο και εγώ υποστηρίζω και φυσικά ο ρόλος μας σαν Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς στην ε, παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου είναι πολύ σημαντική. Το έχουμε τονίσει στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και επίσης στην αμοιβή αναγνώριση επαγγελματικών ε, προσόντων και στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Είναι σημαντικό λοιπόν <clears throat> ότι Πολλές φορές τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην εφαρμογή προέρχονται από την αρχική νομοθεσία και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είτε ότι θέλω να κάνω και μια πρόσκληση προς την Επιτροπή ώστε προτού ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβιάση να δούμε αν υπάρχουν κάποια άλλα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιο επωφέλη. Παραγματικά να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές προς τις κατώτερες ε, αρχές που να διασαφηνίζουν ορισμένα πράγματα ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές ε, διαδικασίες επί παραβιάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μάγια. Πιστεύω ότι έχει συνταχθεί πολύ λογικά και θετικά αυτή η γνωμοδότηση. Νομίζω ότι ένα σημείο που είναι πολύ ενδιαφέρον για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είναι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τις αρχές προς τους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, η, οδηγία για τις μικροδιαφορές, την επίλυση των μικροδιαφορών. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφορές μέχρι 2.000 ευρώ. Κανείς δεν το ξέρει, ούτε καν οι δικαστές παρά το γεγονό ότι θα έπρεπε να έχουν ήδη έντυπα και τα οποία αφορούν την υποβολή τέτοιων διαδικασιών, ούτε και αυτό το γνωρίζουν. Και δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν επίσης ότι υπάρχει κάποια διαδικασία και κάποια προθεσμία για την υποβολή αξιώσεων από επιβάτες, παραδείγματος χάρη αυτοί, αυτοί οι επιβάτες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν λόγω της τέφρας. στην περίπτωση που ξέρω, ένας Γερμανός θέλει να διεκδικήσει 2.000 ε, ευρώ, έχει μια διαφορά με μια Ολλανδική αεροπορική εταιρεία και φυσικά πολλές, πολλές φορές τα δικαστικά, το δικαστικό κόστος υπερκαλύπτει, καλύπτει, υπερκαλύπτει τα λεφτά τα οποία μπορεί να ανακτήσει ο, ο ενδιαφερόμενος. Τώρα, υπάρχει ίσως η δυνατότητα αν υπήρχε δυνατότητα να στραφεί κατά τις εταιρείες η οποία έχει και μια γερμανική, μια ε, γερμανική θηγατρική, αυτό θα ήταν πιο εύκολο γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μονάχα το γερμανικό δικαίωμα. Επομένως, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο πολίτης ποιες είναι οι δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχει. Αν δεν το κάνουν αυτό και τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ασκήσει την απαραίτητη πίεση σε όλα τα κράτη-μέλη για να παρέχουν τις πληροφορίες στους πολίτες. Και εδώ το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και πάλι θέλω να συγχαρώ τον συγγενή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια γιατί ήμουν και εγώ σκιώδης εισηγητής. Αυτό που είναι σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή ειδικότερα είναι ότι είναι πρώτη φορά που συντάσσουμε μια γνωμοδότηση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρονται και θέματα που αφορούν την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες ε, που θεωρούνται σημαντικά ε, σε αυτή την έκθεση και έχει δίκιο ο εισηγητή που τονίζει κάποιε λεπτομέρειε. Ο κύριος Τσαρκόφσκι εξέφρασε κάποιε ανησυχίε, Πάντως εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση έχει πολλά παραδείγματα από συγκεκριμένη νομολογία που δείχνουν ακριβώ αυτό το οποίο κάνουμε. Και το βαθμολόγιο τη εσωτερική αγορά επίση αναφέρεται συγκεκριμένα ω εργαλείο παρακολούθηση. Ένα από τα σχόλια που προκύπτει από προηγούμενες συζητήσεις για το βαθμολόγιο στην εσωτερική αγορά και ίσως θέλουμε να το βάλουμε και στην τελική μας έκθεση είναι το ότι τώρα το έλλειμμα ενσωμάτωσης νομοθεσίας σε εσωτερικό δίκαιο έχει μειωθεί και τα στατιστικά στοιχεία δεν έχουν τόση αποκαλυπτική σημασία. Αυτό που είπε ο Χάνς Πέτερ Μέγερ είναι νομίζω πιο σημαντικό, δηλαδή η πρακτική επίπτωση της νομοθεσίας για τους πολίτες, γιατί μπορεί κάποιο κράτος μέλος να έχει καλά, καλές επιδόσεις στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας, αλλά αν δεν εφαρμόζεται στην πράξη από τους πολίτες αυτό το οποίο έχουμε ψηφίσει, δεν έχουμε καταφέρει και πολλά πράγματα. Αυτή η διαφορά λοιπόν μεταξύ των τυπικών εκθέσεων που εμείς καταρτίζουμε και της εφαρμογής της νομοθεσίας στην πράξη βρίσκεται στην καρδιά αυτής της ε, έκθεσης. Εργαλεία όπως η η αξιολόγηση από ομοτήμους είναι πάρα πολύ χρήσιμα ε, γιατί ε, η επίπτωση, ο αντίκτυπος τη ενσωμάτωση τη νομοθεσία είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι στα κράτη-μέλη και η Επιτροπή οφείλει να ρυθμίζει αυτή τη διαδικασία και να την καθοδηγεί, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δίνει στου πολίτε και κάποιου μηχανισμού ε, εφαρμογή στην πράξη, ούτω ώστε να έχει στην πράξη αντίκτυπο αυτή η νομοθεσία. Και χρειάζεται και στο Κοινοβούλιο να γίνεται περισσότερη δουλειά επ' αυτού. Και σε μία τροπολογία στην έκθεσή σας υπάρχει ακριβώς αυτή η πρόταση, γιατί νομίζω ότι ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει περισσότεροι βουλευτές να ασχολούνται με τα θέματα ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στην Εθνική Νομοθεσία. Όταν κάναμε τη διακοινοβουλευτική συνάντηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες δεν είχαμε τόσο καλή υποστήριξη από τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών και κάποιοι από τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων μας είπαν ότι ότι δεν είχαν ασχοληθεί άμεσα στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτρο στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε και παράλληλα με τις άλλες προτάσεις που έχετε κάνει και αυτή η τροπολογία νομίζω ότι θα βοηθήσει και σας ευχαριστώ για τη γενικότερη αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπο της Επιτροπής εδώ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κρίστιαν ε, Πουζόη, να σας δώσουμε το λόγο για να συνοψίσετε και να κλείσετε αυτή τη συζήτηση και να επιβεβαιώσουμε και το τελικό χρονοδιάγραμμα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές για τις παρατηρήσεις που έκαναν και τις προτάσεις βελτίωσης του κειμένου μου. Όντως υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όπως σας είπα, θα πρέπει η έκθεση αυτή να σεβαστεί πολλά κριτήρια, αν θέλετε. Και έχω προετοιμάσει κάποιες τροπολογίες, τις οποίες έχω διαβιβάσει και στους σκιώδεις συγητές. Τώρα περιμένω και άλλες τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ράπτη. Δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε όσον αφορά τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Επίσης συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Τσαρκόφσκι ότι θα πρέπει να βρούμε έναν πιο ουδέτερο τρόπο για να εκφράσουμε κάποια πράγματα. Δεν έχω αναλάβει πολλές εκθέσεις, οφείλω να ομολογήσω, αλλά οι περισσότερες όμως, για να μην πω όλες οι εκθέσεις μου, ψηφίστηκαν ομόφωνα. Γι' αυτό δεν θα α, τσιγκουνευτώ τις προσπάθειες για να βελτιώσω να τον περισσότερο την έκθεση. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερους κανονισμούς και λιγότερες οδηγίες όσον αφορά το, τη γενικότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν το λέω εδώ, δεν το λέω στην γνωμοδότησή μου, διότι θέλω να την υποστηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Κυρία Ρούλε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα συνδέονται και με τον τρόπο με τον οποίο ε, διατυπώνονται τα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσουμε αν θέλετε αυτούς τους ε, πίνακες ε, αντιστοιχίας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε κάπως και την δουλειά του, των εθνικών κοινοβουλίων. Έχει δίκιο και ο κύριος Μάγερ όταν λέει ότι η πληροφόρηση είναι ζωτική σημασίας. Πληροφόρηση σχετικά με την νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί. Διότι πολλές φορές οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να επωφεληθούν από την νομοθεσία αυτή διότι δεν τη γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ξέρετε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε, στις 4 που θα εξετάσουμε και τις τροπολογίες και την, θα γίνει και η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουζόη. Νομίζω ότι όντως είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά σας, πολύ σημαντικό έργο και θα πρέπει και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να υπερασπιστούμε και τις ε, ε, τροπολογίες μας. Και ο κύριος Μέγερ που ήταν εδώ προηγουμένως θα μας υποστηρίξει. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο που προβλέπεται για την σημερινή μας ε, συζήτηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι η έκθεση του κυρίου Ζουβά, τον οποίο καλωσορίζω είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία της Επιτροπής μας για τι συνέπειε της διαφήμιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών και ε, για τους επισκέπτες μας από το ε, Κολέγιο της Ευρώπης ε, να εξηγήσω ότι οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλία είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να ευαισθητοποιούμε τον περίγυρό μας, αν θέλετε, σε κάποια θέματα. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τις εκθέσεις αυτές, δύο πρωτοβουλίες και θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ο κύριος Ζουβά ε, θα έχει συντάξει την έκθεσή του, την οποία θα ψηφίσουμε το φθινόπωρο η σύνταξη της έκθεσης είναι εν εξελίξη τέλος πάντων. Έχετε νομίζω ότι στη διάθεσή σας αυτά τα έντυπα ε, τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Ε, αναφερόμαστε στις αθέμητες πρακτικές, στις παραπλανητικές διαφημίσεις, ε, θέματα ζωτικής σημασίας για την Επιτροπή μας, ε, γιατί εμείς είμαστε και η, η, αρμόδια καθήλυν Επιτροπή, αν θέλετε, για την οδηγία σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ε, καταρχάς να ρωτήσω τον εισηγητή, θέλετε να παρουσιάσετε τις μελέτες, ε, κύριο Ζουβά, ε, θα πάρετε το λόγο τώρα ή να προχωρήσουμε στην παρουσίαση και θα πάρετε το λόγο μετά. Λοιπόν, απευθύνομαι εδώ τώρα στους εμπειρογνώμονές μας που βρίσκονται εδώ αριστερά. Η κυρία Χάζενχόφε από το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ στο του Βερολίνου, είναι, εδώ είναι όλοι οι, οι συγγραφείς των μελετών. Είσαστε υπεύθυνοι, αλλά έχουμε και τον καθηγητή κύριο Γιάνν Κάμπελ, ε, ομόρφος καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και επίσης ε, έχουμε τον δόκτορα Φρανκ Άλεβελτ, ο οποίος είναι υπεύθυνος, ανέλαβε μάλλον τη σύνταξη της έκθεσης και ξέρω ότι έχετε κάνει ε, ως ανυπεργολαβία και έχει κάνει ε, πολλές εκθέσεις και για τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Σας καλωσορίζω όλους θερμά. Έχουμε τις διαφάνειες ε, τις οποίες βλέπετε στις οθόνες. Η καθηγήτρια κυρία Σουζάννα Χάουγενχόφερ ε, θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ με προσκαλέσατε να παρουσιάσω τα κύρια πορίσματα της έρευνάς μας. Το θέμα μας ήταν η κατάσταση εφαρμογής της, των διατάξεων της νομοθεσίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην περίπτωση της διαφήμισης και επίσης τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Η δομή της παρουσίασης έγινε με ερωτηματολόγια, με συνεντεύξεις με τους ε, εμπλεκόμενους σε έξι Η δομή της παρουσίασής μου είναι η εξής. Καταρχήν το UCPD, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές δηλαδή, η κατάσταση εφαρμογής, τα προβλήματα εφαρμογής και αστυνόμευσης και ο ρόλος των ρυθμιστικών φορέων για την διαφήμιση. Θα δούμε τα θέματα αυτά πρώτα από μια γενική προσέγγιση και μετά θα εστιάσουμε στις αθέμητες πρακτικές παραπλανητικής διαφήμισης στο ίντερνετ. Η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ενεκρίθη το Μάιο του 2005 και θα έπρεπε Μπορείτε να πάτε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι το, τις 12 Ιουνίου του 2007. Ορισμένα μέλη όμως, μεταξύ των οποίων η Φιλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθυστέρησαν στην εφαρμογή αυτής τη οδηγία. Σήμερα βέβαια όλα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση του δικαίου για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που μπορεί να θίξουν τα οικονομικά συμφέροντα των ε, καταναλωτών μεταξύ των οποίων και η παραπλανητική διαφήμιση που θα μπορούσε να δημιουργήσει ασάφειες, αβεβαιότητες και να παραπλανήσει τους ε, καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο σημαντικές ε, πτυχές όπου φαίνεται υπερ, τα όρια της οδηγίας για την, ε, τις αθέμητες πρακτικές. Αφορούν πρακτικές οι οποίες θίγουν τους καταναλωτές, αλλά δεν αναφέρεται σε θέματα παραγωγής χάρη ε, ηθικής ή αξιοπρέπειας. Αφορούν λοιπόν τις σχέσεις ε, επιχειρήσεων με καταναλωτές και <clears throat> βάσει αυτής της οδηγίας δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυστηρότερη νομοθεσία αλλά η οδηγία αυτή έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Αφορά όλες τις ε, μεμονωμένες ενέργειες σε περίπτωση που προκύπτει κάποια ζημία για καταναλωτές, αλλά δεν πάντα με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για το συμβατικό δίκαιο και, την, ε, και τις αποζημιώσεις έχει ένα γενικό, μια γενική ρήτρα, το άρθρο 5, και δύο μικρότερες ρήτρες που είναι οι παραπλανητικές πρακτικές και οι επιθετικές πρακτικές. Οι δύο αυτές τελευταίες ρήτρες απαγορεύουν τις παραπλανητικές ε, και επιθετικές εμπορικές διαδικασίες. Και η γενική ρήτρα είναι το δίκτυο ασφαλείας και εφαρμόζεται μονάχα εάν δεν καλύπτεται από το, αν δεν καλύπτεται από το παράτημα 1, τη μαύρη λίστα ή οποιαδήποτε άλλη από τις δύο προηγουμένως αναφερθήσεις ε, ειδικέ ρήτρε. Τα κάτι μελη πρέπει να απαντήσουν σε δύο βασικά ερωτήματα για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Πώς, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμοστεί και πώς. κάτι <clears throat> κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την οδηγία μέσα στην κωδικοποίηση που έχουν, παραγωγή χάρη, στις νομοθετικές πράξεις κατά του του ανταγωνισμού, στον κώδικα ε, καταναλωτή ή σε άλλες, σε άλλα νομοθετικά μέτρα ή στο αστικό δίκαιο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει καλυφθεί με, κάποια, με κάποιο κανονισμό ο οποίος μεταφέρει την οδηγία αυτή. Όπως είπα, αφορά αυτή η οδηγία μονάχα εμπορικές πρακτικές από οδηγια μοναχα εμπορικες πρακτικες απο επιχειρησει προς καταναλωτές κάποια κράτη-μέλη, αλλά όχι όλα, <clears throat> έχουν εφαρμόσει με αυτή τη στενή ερμηνεία την οδηγία αυτή. Αλλά δεν είναι σαφές από την εφαρμογή ότι αφορά μονάχα τις σχέσεις επιχείρησεων προς καταναλωτές. Στη Γαλλία εφαρμόστηκε στον κώδικα καταναλωτή, αλλά οι, οι διατάξεις για την παραπλανητική διαφήμιση αφορούν επίσης και σχέσεις μεταξύ επιχείρησεων, B2B. Ας δούμε λοιπόν τώρα το θέμα των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Οι πρακτικές αυτές καλύπτονται από την οδηγία αυτή, ιδιαίτερα στο άρθρο 2, όπου αναφέρονται οι εμπορικές πρακτικές ως οι παραπλανητικές πρακτικές ως οποιαδήποτε πράξη παράληψης ή διατύπωσης σε σχέση με τα θέματα αυτά από τους εμπόρους οι οποίοι συνδέονται απόλυτα με την πρόθεση ενός προϊόντος προς τον καταναλωτή. Είναι παραπλανητικές πράξεις ή παραλήψεις. το άρθρο 6 αφορά τις παραπλανητικές πράξεις, το 7 τις παραλήψεις ή επίσης υπάρχει γενική ρήτρα του άρθρου 5 η οποία μπορεί να καλύψει τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το άρθρο 1 <clears throat> αναφέρεται σε 23 μορφές παραπλανητικών πρακτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση του καταναλωτή η οδηγία ε, απαγορεύει τόσο την ψευδή όσο την αληθή αλλά και παραπλαντική πληροφόρηση στον ίντερνετ που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Αλλά το ίντερνετ υπόκειται σε γρήγορες μεταλλαγές που επηρεάζουν και τις τεχνικές μάρκετινγκ είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις και τις νομικές τους συνέπειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια τελική κρίση για το αν η οδηγία για τις καταχρηστικές προ... πρακτικές είναι επαρκής για να καλύψει όλες αυτές τις αναδυόμενες πρακτικές. Αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι παρά τις ιδιαιτερότητές τους οι παραπλανητικές διαφημίσεις στο ίντερνετ θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες νομικές προδιαγραφές όπως και οι άλλες μορφές διαφήμισης. Μια διαφήμιση που λέει ότι όλα τα προϊόντα που αναφέρονται είναι προς πώληση, αλλά κάποια από αυτά δεν είναι, αυτό είναι μια παραπλανητική ε, διαφήμιση. Θα αναφερθώ τώρα σε τρεις κατηγορίες παραπλανητικών διαφημίσεων στο ίντερνετ. Υπάρχουν οι εξής τάσεις σε σχέση με τις παραπλανητικές, με τα ε, πρακτικές αυτές. Καταρχήν υπάρχουν οι ενκρυπτό διαφημίσεις στο ίντερνετ που δεν αποκαλύπτουν στον ε, καταναλωτή την εμπορική μορφή αυτής της δράσης. Παραδείγματο χάρη περιγραφές ή κριτικές προϊόντων όπου φαίνονται κάποιοι οι οποίοι γράφουν σαν καταναλωτές αλλά στην πραγματικότητα έχουν πληρωθεί από τους παραγωγούς αυτού του προϊόντος. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή νομικέ αποφάσει, δικαστικέ αποφάσει για τα θέματα αυτά. Αυτή η μορφή εν κρυπτό, δηλαδή διαφήμιση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί. Ακόμα και αν φαίνεται ύποπτη μία παρουσίαση ενό προϊόντο, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει κανεί ότι αυτό ο οποίο έγραψε αυτή την παρουσίαση πράγματι ή το αργυρώνητο είχε πληρωθεί από τον παραγωγό του προϊόντο. Επίσης, Πολλές φορές τα δίκτυα κοινωνικής επαφής δίνουν την εντύπωση ότι έχουν επιλεγεί κάποια άτομα επειδή έχουν παραγωγός καλή εμφάνιση και μπορούν να προωθηθούν σε μια καριέρα μοντέλου. Και με τον τρόπο αυτό αποσπώνται πληρωμές, μικροπληρωμές. Άλλη μορφή τέτοιας παραπλανητικής διαφήμισης στο ίντερνετ είναι η διαφήμιση με σήματα ποιότητας. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες μορφές που μπορούν να διακριβωθούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ε, σήματα ποιότητας τα οποία δεν είναι, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτή η επιχείρηση. Η δεύτερη ομάδα περιπτώσεων είναι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ε, πεπαλαιωμένες ή ε, πεπαλαιωμένα σήματα ή σήματα ποιότητας που έχουν εκπνεύσει σε σχέση με την χρονική τους ισχύ. Τρίτη περίπτωση είναι περιπτώσεις οποίες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήματα τα οποία δημιουργούν την εντύπωση ότι εκπληρούν κάποιες ειδικέ προδιαγραφές ποιότητος και γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτά τα σήματα. Αλλά στην περίπτωση αυτή η ετικέτα αυτή απαιτεί μονάχα ορισμένε νομικές διαδικασίες και όχι διαδικασίες ποιότητας. Επομένως είναι παραπλανητική στην περίπτωση αυτή. Παραγωγός χάρη σε σχέση με την φροντίδα που πρέπει να ασκήσει ο παραγωγός σε σχέση με το προϊόν. Φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις παραπλανητικής διαφήμισης στο ίντερνετ ε, μεγάλο μέρος παίζουν ε, οι ασφαλμένες ε, παραπλανητικές τιμές που αναγράφονται. Και εδώ έχουμε τρεις περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε περιπτώσεις όπου η τιμή η οποία αναφέρεται στο ίντερνετ είναι παραπλανητική διότι δεν αναγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής ανακαλύπτει ο καταναλωτής συμπληρωματικές ε, επιβαρύνσεις μόνο αφού πατήσει το κουμπί. Τέτοιες πρακτικές έχουν αναφερθεί ιδίως ε, για αεροπορικά εισιτήρια και για διάφορες συμβάσεις Παραδείγματος χάρη όταν μια τιμή προσφέρεται ε, για συγκεκριμένη περίοδο και όχι για τη συνολική περίοδο διαμονής σε ένα ξενοδοχείο παραδείγματος χάρη. Δεύτερη περίπτωση είναι όταν ε, υπάρχει μια προσφορά που αναφέρεται ως δωρεάν και ε, εδώ έχουμε πολλά περιστατικά υπηρεσιών που παρέχονται. Παραδείγματο χάρη ε, για το κατέβασμα μουσική ή για την αποστολή μηνυμάτων ή για το οροσκόπιο που διαφημίζονται ω δωρεάν υπηρεσίε στο ίντερνετ. Ο καταναλωτής όμως θα πρέπει να συμπληρώσει κάποιες προσωπικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα για να μπορέσει να λάβει την υπηρεσία και μόνο αφού εγγραφεί και αφού πάρει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι ε, μια σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ε, συμπεριλαμβανόταν σε αυτό το οποίο ζήτησε και συνήθως οι πληροφορίες για τη σύναψη της σύμβασης δίδονται μόνο αφού έχει δώσει προσωπικά δεδομένα ο καταναλωτής. Επιπλέον, οι πληροφορίες δίνονται με πολύ μικρούς χαρακτήρες δυσανάγνωστους και ο καταναλωτής μαθαίνει για τη σύμβαση μόνο αφού του σταλεί το τιμολόγιο και κάποιος δικηγόρος έρχεται σε επαφή με τους ε, καταναλωτές. Είναι επιθετική λοιπόν η συμπεριφορά των ε, εταιριών που προσπαθούν να ζητήσουν τα χρήματα από τους καταναλωτές. Ε, τελευταία κατηγορία αφορά τις συγκρίσεις τιμών. Ιστότοποι με συγκρίσεις τιμών μπορεί να περιλαμβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες. Δεν αναγράφονται ορισμένες φορές ε, οι πραγματικές τιμές των ε, αεροπορικών εισιτηρίων ε, για κάποιες ε, προσφορές και δεν ενημερώνονται οι καταναλωτές για όλες τις λεπτομέρειες. Δεύτερον, οι συγκρίσεις τιμών θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Μια διαφήμιση που συγκρίνει τιμές τηλεφώνων θα έπρεπε να ενημερώνει και για την ελάχιστη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης. Μια διαφήμιση που λέει ότι η τιμή είναι χαμηλότερη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες για τη συνολική τιμή. Τώρα, περνάμε στα προβλήματα και τις δυσκολίες της ε, εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ των ερωτωμένων υπήρχε συμφωνία ότι υπάρχει ασάφεια, νομική ασάφεια για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Η ασάφεια και η αβεβαιότητα ίσως ε, οφείλεται σε αόριστες διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται στις γενικές ρήτρες της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Κατά τη γνώμη πολλών εμπλεκομένων, αρνητικός κατάλογος που συμπεριλαμβάνεται, αυτό το black που συμπεριλαμβάνεται, δεν έχει αρκετά πληροφοριακά στοιχεία για να ερμηνευθεί σωστά και δεν τηρούνται και οι απαιτήσει του παραρτήματος 1 για τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση, Ιδίως το άρθρο 7 της οδηγίας μπορεί να δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές επηρεάζεται και από θέματα προσωπικής ε, επιλογής ή αξιοπρέπειας, παρότι δεν καλύπτονται αυτά τα θέματα. Και τα πρότυπα ε, αξιοπρέπειας ε, και προσωπικής επιθυμίας μπορεί να επικύλουν από το ένα κράτος μέλος ε, στο άλλο. Για να μην υπάρχει αβεβαιότητα, λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφώς είναι χρήσιμες, Κάποια κράτη δίνουν κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουν και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αυτές οι εθνικές κατευθυντήριες αρχές μπορούν να βοηθήσουν διότι εξασφαλίζουν ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη αλλά δεν συνεισφέρουν σε ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή μια επίσημη βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει αποφάσεις από τα εθνικά δικαστήρια και από φορείς επιβολής της νομοθεσίας ε, στην αγγλική γλώσσα, διαθέσιμη προς όλους, θα είναι σημαντικό μέτρο για να τονίσουμε την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας. Μια τέτοια βάση δεδομένων διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο του 2010. Επιπλέον, η έκδοση περαιτέρω κατευθυντηρίων γραμμών για την ερμηνεία της οδηγίας για τις αθέμητε εμπορικές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα μέτρο το οποίο είναι προ σκέψη και η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί διαφορετικά εκτό ε, ε, εάν ε, ληφθούν πολλές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ρήτρα για την πλήρη εναρμόνιση απαιτεί από τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν το εθνικό τους δίκαιο προς την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και να αποφύγουν διαφοροποίησεις από τα πρότυπα τα οποία θεσπίζει η οδηγία. Η διαδικασία υλοποίησης επομένως απαιτεί όχι μόνο την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και την τροποποίηση ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας εάν παραβιάζει την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές παραμένει προ διερεύνηση το αν έχουν επιτύχει τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αντιμετωπίσει τρία προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ε, μη έγκριση, με μη εφαρμογή εθνική νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη για την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχει ακόμη μια ε, εκκρεμούσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απαγόρευση προσφορών σε κάποιο κράτος μέλος και για το αν αυτό παραβιάζει την οδηγία. Η οδηγία προβλέπει πλήρη εναρμόνιση και μόνο οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές του παραρτήματος 1 θεωρούνται αθέμητες ε, ε, ούτως ή άλλως. Όλες οι άλλες εμπορικέ πρακτικές είναι αθέμητε, εάν εμπίπτουν σε μία από τις γενικές ρήτρε. Ίσως ε, ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη έχουν τέτοιες διατάξεις ή παρόμοιε διατάξει στο εθνικό δίκαιο που δεν είναι συμβατές με την οδηγία για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικές λαμβάνοντα υπόψη το καθεστώ τη πλήρου πλήρους Η υπόθεση, η προδικαστική διαδικασία που εκκρεμεί ακόμη μας ε, ε, υποδηλώνει άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει για την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια διαδικασία απαγόρευσης ε, δωρεάν προσφορών από περιοδικά και εφημερίδες που απαγορεύεται στην Αυστρία. Η αυστριακή κυβέρνηση λέγει ότι ο στόχος αυτής της διάταξης στην Αυστρία δεν είναι μόνο η προστασία των καταναλωτών, αλλά και η προστασία των μικρών ανταγωνιστών για να μπορέσει να υπάρχει διαφοροποίηση των τιμών. Η οδηγία δεν αφορά τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Όμως η προστασία των καταναλωτών από αθέμητες εμπορικές πρακτικές ενδέχεται να προστατεύει και τις επιχειρήσεις που ακολουθούν θεμητές πρακτικές. Εφόσον η οδηγία προβάλλει ομοιόμορφες ομοιόμορφη εφαρμογή, δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν αυστηρότερες διατάξεις. Ίσως λοιπόν ε, οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, παραβιάζουν την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μπορούν όμως οι αυστηριακές αρχές να συνεχίσουν να απαγορεύουν αυτή την προσφορά από περιοδικά και εφημερίδες αν δεν εντάσσεται στην οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δηλαδή τελικά μπορεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πιο αυστηρές νομοθεσίες, πιο αυστηρές διατάξεις από ότι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη όταν πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία. Όπως ήδη είπαμε, το άρθρο 3 την υποπαράγραφο ε, 3 λέει ότι δεν ε, ε, φύγεται το δίκαιο των συμβάσεων παράλληλα. Λέγεται ότι αυτό ισχύει στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά μια εμπορική, μια εμπορική συναλλαγή. Θα υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις και στο εθνικό δίκαιο των συμβάσεων, ιδιαίτερα για τις προσυμβασιακές πληροφορίες το άρθρο 7 της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που απαγορεύει τις παραπλανητικές ε, παραλήψεις ε, πληροφόρησης ε, αποτελεί ένα νέο στοιχείο για, πολλά, για πολλές περιπτώσεις δικαίου των συμβάσεων. Εάν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το DCFR, για τη λήψη των κατάλληλων νομικών μέτρων. Όσον αφορά την υλοποίηση τώρα την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, το άρθρο 11 αφήνει διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Τα συστήματα επιβολής νομοθεσίας σε άλλα κράτη-μέλη κυμαίνονται από συστήματα αστικού δικαίου μέχρι διοικητικό δίκαιο και συστήματα που συνδυάζουν και τα δύο. Αυτή η ομάδα των κρατών στηρίζεται ε, σε κυρώσεις ε, που προβλέπει το οστικό δίκαιο και σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να δώσουν τα δικαιώματα στους καταναλωτές να αναθεωρήσουν. Σύμφωνα, παραδείγματο χάρη, με την πράξη της, για την προστασία της, του καταναλωτή της ε, Ιρλανδίας, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Επίσης, ο νόμος που μεταθέτει την οδηγία αυτή ε, επιτρέπει στον καταναλωτή να προσφύγει στα δικαστήρια. Υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές στα εθνικά συστήματα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιες διασυνοριακές ε, συναλλαγές και προβλήματα, διότι πολλές φορές οι καταναλωτές δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Όσον αφορά την συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα συστήματα εφαρμογής, η συνεργασία αυτή προς, για την προστασία των καταναλωτών προσφέρει την απαραίτητη ενημέρωση και συνεργασία. κυρίως όσον αφορά τις διοσυνοριακές, διοσυνοριακή εφαρμογή, υπάρχει κάποιο συντονισμό και συνεργασία, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα κενά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργεί η διαφορετική γλώσσα και εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον ε, παραβιάζεται η οδηγία ή όχι. Ε, τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε για τις προπλανητικές διαφημίσεις στο ίντερνετ είναι το ιδιαίτερο πρόβλημα που, που παρουσιάζουν οι απαταιώνες έμποροι και υπάρχουν πολλές ε, τέτοιου είδους ε, υποθέσεις τις οποίες έχει εξετάσει το, η Υπηρεσία Προσεστού Καταναλωτή στην Γερμανία. Βέβαια, οι κυρώσεις που προβλέπονται δεν ε, εφαρμόζονται ε, επαρκώς. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ε, στο ίντερνετ μπορεί να κλείσει το ένα site και να ανοίξει κάποιο άλλο αυτός ο απαταιώνας, αν θέλετε. η γερμανική νομοθεσία μπορεί θεωρητικά να είναι χρήσιμη, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει στεφθεί με επιτυχία. Για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τους απαταιώνες, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές ποινές, πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Τώρα, όσον αφορά την αυτορύθμιση, το άρθρο 10 της Οδηγίας για τις Αθέμητες Εμπορικές Πρακτικές ε, προβλέπει τέτοιου είδους δυνατότητες αυτορύθμισης είναι το σύστημα της συνύπαρξης αν θέλετε και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ε, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιτρέψουν την αυτορύθμιση των εμπορικών πρακτικών. Η οδηγία αναφέρεται σε κώδικες συμπεριφοράς σε πάρα πολλές περιπτώσεις και απαγορεύει τις παραπλανητικές αναφορές στους κώδικες ε, συμπεριφοράς. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 12, τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν το πόσο θα εφαρμοστεί η, οδηγία. Και η αυτορύθμιση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την μετάφορά της και την εφαρμογή της οδηγίας. Η σημασία των εθνικών σωμάτων ή υπηρεσιών αυτορύθμισης ε, διαφέρει από κράτος μέλους σε άλλο. Όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση στο ίντερνετ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι όλα όλοι οι κώδικες ε, αυτό, ε, δεν συμπεριλαμβάνουν τέτοιου είδους κώδικες συμπεριφοράς. Ορισμένοι φορείς αυτορύθμισης αφορούν μόνο τα θέματα αξιοπρεπίας, ας πούμε. Αυτό ισχύει για την Αυστρία, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει την παραπλανητική διαφήμιση, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους κώδικες αυτορύθμισης η διαφήμιση πρέπει να είναι ειλικρινής. Και στην Γερμανία αναφέρονται μόνο τα θέματα αξιοπρέπειας. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Ε, εκεί υπάρχει μια, ένας ευρύτερος, ένα ευρύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων που έχουν οι φορεί αυτορύθμιση. Υπάρχουν όμως και κάποιοι περιορισμοί, του οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ε, ο κώδικας αυτορύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν καλύπτει τις ε, διαφημίσεις ε, για τις επιχειρήσεις στο homepage. Επίσης, οι, οι φορείς αυτορύθμισης ε, θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο οι προσπάθειες αυτορύθμισης όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση. Το 2008 ε, μια ένωση για τις ε, διαφημίσεις ε, έχει υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Αναφέρεται παραδείγματο χάρη ε, και τα θέματα της ε, ψηφιακής, ε, των ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών και πόσο μπορούν να ρυθμιστούν με διαδικασίες αυτορύθμισης. Η οι, αυτο, οι φορείς αυτορύθμισης μπορούν να ε, ρυθμίσουν ε, τις απλές περιπτώσεις ε, όσον αφορά τις διαφημίσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό κερδίζουμε και χρόνο και χρήματα. Γι' αυτό και οι κώδικες συμπεριφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα θέματα παραπλανητικής διαφήμισης στο ίντερνετ. θα πρέπει ε, παραδείγματο χάρη να μπορούν να υποβάλλονται παράπονα ελεύθερα και θα πρέπει ε, οι φορείς αυτορύθμισης να μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει αυτοί οι φορείς να είναι ανεξάρτητοι να μην ε, να ε, μπορούν να προβλέψουν απαραίτητες ε, κυρώσεις και ποινές στην επιχειρήση η οποία αρνείται να συνεργαστεί. Αν δεν μπορέσουν οι αρχές αυτών των φορέων αυτορύθμισης να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους στην, στην επιχείρηση, θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν σε ένα ανώτερο όργανο, γιατί, και γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως και η, η Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία προβλέπεται. Σε κάποια κράτη-μέλη αυτά τα συστήματα ήδη έχουν εφαρμοστεί. Βέβαια δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις εμπορικές πρακτικές που καλύπτονται από την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, κυρίως όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παράπονα να υποβάλλονται άμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς αυτορύθμισης. Το σύστημα όμως αυτό δεν μπορεί να <clears throat> λειτουργήσει εφόσον δεν υπάρχει κάποιος κώδικας συμπεριφοράς και εφόσον δεν υπάρχει η θέληση να υπάρχει συνεργασία με τις ρυθμιστικές ασχέσεις. Επομένως ένα σώμα αυτορύθμισης θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το κανόνα. Επίσης οι κώδικες αυτορύθμισης και αυτοπεριορισμού θα πρέπει να έχουν και ένα κώδικα ο οποίος να εφαρμόζει την οδηγία για την, τις ε, αθέμητες πρακτικές και σε σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και να δίνει κατευθυντήριε γραμμέ για τι επιχειρήσει και με τον τρόπο αυτό μπορεί να προωθήσει μια καλύτερη συμμόρφωση με τον κώδικα αυτό και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κυρία, <clears throat> κυρία μου για την τόσο πλήρη έκθεσή σας, η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα. Δεν είναι μονάχα το πλαίσιο της μονάχα, που συνδέεται με την έκθεση του κ. Ζουβέντα, αλλά συνδέεται και με την έκθεση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σίγουρα καταδεικνύεται μερικά από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα σχόλια σας λοιπόν σίγουρα δείχνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν και την ανάγκη εφαρμογής ε, Αυτόν των διατάξουν πολλές φορές και σε σχέση μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε την περίπτωση της Αυστρίας όπου εφαρμόζεται με πιο αυστηρό τρόπο αυτή η νομοθεσία. Η... Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει με την διαδικασία της πλήρους εναρμόνσης. Χάρη στον κύριο Ζουβέντ λοιπόν έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία και τώρα φυσικά έχουμε χρόνο να ακούσουμε την άποψη των μελών της Επιτροπής μας και δεν ξέρω προηγουμένως αν θέλει κάποιος από τους ε, συνεργάτες σας να προσθέσει κάτι ή αν θέλετε απλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα. Θα ακούσουμε τα ερωτήματα. Ωραία. Θα σας δώσω τη δυνατότητα στο τέλος να απαντήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας να κάνει κάποια σχόλια εφόσον το επιθυμεί. Ίσως έχει να κάνει κάποια πρόσθετα σχόλια σε σχέση με την παρουσίασή σας και όποιοι άλλοι θέλουν να λάβουν το λόγο Επίσης, ο κύριος ε, Ζουβέν, η κυρία Ρούλε, επίσης η κυρία Στάιλερ. Κύριε Ζουβέν, έχετε πρώτο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτού του σημειώματος αυτής της έρευνας για την ποιότητα της εργασίας τους. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα και έχω να θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα αυτορύθμιση. Εθελοντική ρύθμιση. Λέτε ότι αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλα τα κάτι μελη αλλά τα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου, ίσως δεν είναι επακριβή και θέλω να έχω την απόψή σας, δείχνουν ότι ορισμένα κράτη-μέλη <clears throat> δεν έχουν ακόμα φορείς εθελοντικής ρύθμισης, όπως είναι η Κύπρος, η Μάλτα, η Εστονία, η Λετωνία. Μου λένε ότι στην Δανία μόλις ξεκινάει η λειτουργία ενός τέτοιου φορέα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα λοιπόν, γιατί είπατε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν φορείς αυτορύθμισης. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Δεύτερο ερώτημα. Εδώ θέλω να θέσω το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ καταναλωτών, του, όχι μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, αλλά μεταξύ καταναλωτών βλέπουμε στο ίντερνετ να υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη δραστηριότητα συζητήσεων για όλα τα θέματα. Και οι εταιρείε σήμερα υπόκεινται ιδιαίτερα στους κινδύνους από την διάδοση φημών. Η εταιρεία Περιέ που παράγει το γνωστό εμφιαλωμένο ε, χρειάστηκε να αποσύρει χιλιάδες φιαλών και αυτό οδήγησε σε πτώση της, ε, της μετοχής του, της εταιρείας αυτής στα χρηματιστήρια, γιατί κυκλοφόρησε μια φήμη ότι είχε γεύση πετρελαίου, ότι ορισμένες παρτίδες του προϊόντος αυτού είχαν γεύση πετρελαίου. Επομένως, τίθεται το θέμα αυτό του να βρούμε μια νέα μορφή, να καθορίσουμε τι ακριβώς είναι η διαφήμιση άμα βγω εγώ και πω ότι το εστιατόριό σας είναι πραγματικά άχρηστο, είναι πολύ κακής ποιότητος και κάποιοι φίλοι μου κάνουν το ίδιο πράγμα, μπορούμε να κάνουμε ένα είδος αντιδιαφήμισης, αρνητικής διαφήμισης, το οποίο μπορεί τελικά να οδηγήσει σε βλάβες για τις επιχειρήσεις, σε ζημίες στις επιχειρήσεις και να θίξει το δικαίωμα του επιχειρήν. Επίσης για την οδηγία για τις ε, αθέμητες πρακτικές. Κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται να λειτουργεί ιδιαίτερα καλά είναι η σχέση μεταξύ κρατών. Εάν εγώ καταθέσω μια αγωγή εναντίον ενός παραγωγού ή ενός διανομέα σε ένα άλλο κράτος μέλος, τα πράγματα μπερδεύονται ήδη από την αρχή. Γιατί πρέπει αυτή η αγωγή να εκδικαστεί καταρχήν σε εθνικό επίπεδο στο δικό μου κράτος και μετά να ε, διαβιβαστεί σε μια διοικητική αρχή σε ένα άλλο κράτος όπου βρίσκεται αυτός ο οποίος μου πούλησε αυτό το προϊόν και ξέρουμε ότι αυτά δεν λειτουργούν πολύ καλά. Υπάρχει ένας κανονισμός για διοικητική αρρωγή, ο οποίος υπάρχει ήδη. Είναι ο κανονισμός 2004-2006, όπως λέμε στην αργό μας. Αλλά η εσωτερική αγορά δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει την απόλυτα καλή λειτουργία τέτοιου είδους αγωγών που είναι διαμεθοριακού χαρακτήρα. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας λοιπόν σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρούιλε, κυρία Τέρνερ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Δεν το διάβασα ακόμη το κείμενό σας, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση για μας που παρακολουθούμε τα θέματα της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και είδα και πολλά σημεία που έχουν άμεση σχέση. Μια ερώτηση που έχει σχέση με τη σελίδα 13 για την πλήρη εναρμόνιση. Αυτό το blacklist έχω ακούσει ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρω αν έχετε παραδείγματα σχετικά. Εγώ έχω τουλάχιστον ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. Εδώ και χρόνια έχουμε μια απαγόρευση για τα κουπόνια εκτόσεων. Όλα τα πολιτικά κόμματα αποφάσισαν ότι είναι κάτι το ανεπιθύμητο και θέλουμε να σταματήσουμε να υπάρχουν προς όφελος των καταναλωτών μας. Χάρη στο blacklist, επειδή δεν είναι στο blacklist, δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτή την απαγόρευση. Και αυτό εγώ το θεωρώ πρόβλημα, μπορείτε να το σχολιάσετε. Δεν ξέρω αν εξετάζετε με μονομένα εθνικά παραδείγματα, αλλά κάποια σχόλια και για αυτά τα εθνικά παραδείγματα θα ήταν χρήσιμα. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε κυρία Τούρνεν, η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίασή σας δείχνει πόσες πολλές διαφορές υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στην ε, Σκοτία ε, νομίζω ότι θα θύμωναν πάρα πολύ ε, εκλογής μας αν τους απαγορεύαμε τα κουπόνια, τα εκπτωτικά από τις εφημερίδες. Για το σημείο που αναφέρεται για τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, ένα θέμα είναι αυτοί οι οδηγοί πόλεων που υπάρχουν. Αν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις σε αυτούς τους καταλόγους, ε, σε αυτούς τους οδηγούς ε, πόλεων. Ε, είδαμε πολλά θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Υπάρχουν sites όπως το eBay και άλλα, στα οποία οι καταναλωτές προσφέρουν για αγορές. Και σίγουρα μας ενδιαφέρουν οι διαφημίσεις αυτές τις ιστοσελίδες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση γιατί μας έδωσε πολλά να σκεφτούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Στάιλερ από τη συζήτηση για την οδηγία περί πρακτικών, εμπορικών πρακτικών, θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι δεν θέλαμε να κάνουμε πολύ, πολύ πλοκή αυτή τη συζήτηση και φαίνεται ότι οι αυστριακές αρχές ε, κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο ε, εμεί θέλαμε να αποφύγουμε, αλλά μάλλον ε, είναι υπερβολικά, δείχνουν υπερβολικό ενθουσιασμό, υπερβολικό ζήλο οι Αυστριακέ αρχέ. Η κυρία Κράτσα Μπίλ. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν παιδιά θα έχετε ζήσει ε, την μάχη ε, για να πάρεις που θέλουν τα παιδιά να αγοράσουν οδοντόκρεμα που έχει Mickey Mouse, τα κόνφλεξ που έχουν κάτι άλλο και ανάμεσα στη μάχη που πρέπει να δώσεις ε, και να έχεις την ησυχία σου, ε, οι περισσότεροι αγοράζουν τα προϊόντα. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Άρα σε αυτή την τόσο εξαιρετική δουλειά που κάνει ο φίλος μας ο Φιλίπ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα των πλέον ευάλωτων και πιο εύκολα χειραγωγήσιμων ε, πολιτών μας που είναι τα παιδιά. Θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Τη μελέτη τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για την εφαρμογή. Το πρόβλημα για την ελάχιστη εναρμόνιση είναι το κατά πόσο μπορούν να το εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Δεν με εκπλήσουν λοιπόν εδώ αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά ε, είδα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το έχουν μεταφέρει ως κανονισμό και στην Αυστρία και στη Γερμανία ε, έχει ενταχθεί στο σύστημα ε, αντιμετώπισης των επιχειρήσεων και δεν είναι τόσο σαφές το ποια επίπτωση έχει αυτό για τους καταναλωτές στην κάθε χώρα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί θεωρείτε πιο αποτελεσματική την εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη γνώμη σας. Um, θα ήθελε κανείς άλλος να πάρει το λόγο ε, σε αυτόν τον πρώτο γύρο, ο κύριος Τσαρκόφσκι. Μία πάρα πολύ σύντομη ερώτηση για αυτή την σύγχυση που υπάρχει ανάμεσα στους έμπορους και στις επιχειρήσεις στο ίντερνετ και κυρίως όσον αφορά τους πληστηριασμούς τους online πληστηριασμούς τι είναι παραπλανητικό ας πούμε για τους καταναλωτές όταν μια επιχείρηση φαίνεται ότι είναι ένας έμπορος ο οποίος πουλάει μεταχειρισμένα είδη και προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι φοβερή ευκαιρία, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι το προϊόν του. Διότι πολλές φορές ε, υπάρχει, ε, υπάρχουν ασαφή όρια ανάμεσα στους, ε, στους επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και τους εμπόρους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος πριν ζητήσω από τους εμπειρογνώμονές μας ε, να μας ε, να απαντήσουν, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω διάφορα άτομα. Καταρχάς, τον κύριο Μόντι, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά για τις αθέμητες διαφημίσεις. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω και την αντιπροσωπεία από το EMP ΤΕ της, τη Γαλλία που ήρθαν εδώ για να ακούσουν ε, την ε, παρουσίαση του κυρίου Ζουδά. Σας καλωσορίζουμε όλους και τώρα χαίρομαι που μπορώ να δώσω το λόγο στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων μας. Δεν να πάρει το λόγο. Η καθηγήτρια κυρία Άγγενχόφερ ίσως και μετά θα ζητήσουμε και από τους συναδέλφους σας να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να διευκρινίσω κάτι. Καταρχάς να απαντήσω για την, προτελευταία εναρμόνιση, πρόκειται για... η προ... ερώτηση, πρόκειται για πλήρη εναρμόνιση και όχι μερική. Επίσης δεν είπα ότι η μεταφορά της, στο Ηνωμένο Βασίλειο της οδηγίας έχει γίνει είναι καλύτερη από ό,τι στην Αυστρία ή στη Γερμανία. η οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Τώρα από εκεί και πέρα πώς θα γίνει αυτό, πώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, είναι θέμα εθνικό αν θέλετε. Τώρα, για να επανέλθω στην πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά την αυτορύθμιση. Σύμφωνα με την, ε, οργάνωση, την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ομπρέλα, Υπάρχουν σώματα αυτορύθμισης σε όλα τα κράτη, αλλά δεν μπορούσα να, δεν μπορούσα να στείλω ρευματολόγιο και στα 27 κράτη-μέλη. Άρα πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω στην Εστονία, στην Μάλτα ή στην ε, Δανία πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά όσο πιο ανεπτυγμένη η νομοθεσία για, την, για, τον, για την, αθέμητο ανταγωνισμό, τόσο πιο εύκολη είναι η λειτουργία των φορέων αυτορύθμισης. Γι' αυτό η, Γι' αυτό σε ορισμένα κράτη όπου τα θέματα αθέμη του ανταγωνισμού ρυθμίζονται από τις αρχές του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά φαντάζομαι. Θα ήθελα να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Ερώτηση που έθεσε ο κύριος Σουζουζά. Για την, ε, περίπτωση, για την υπόθεση Περγέ είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα μέσα στα πλαίσια της οδηγίας αθέμη των εμπορικών πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ρύθμισε την, έλαβε την απόφασή του με βάση το άρθρο 10 για τη Σύμβαση, τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναφέρθηκε και στο δικαίωμα αρνητικών σχολείων εις βάρος μιας άλλης επιχείρησης. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μας προσφέρει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Επομένω, αυτού του είδους τα αρνητικά σχόλια, τα επικριτικά σχόλια τα οποία κάνουν, μπορούν να κάνουν ιδιώτες, δεν καλύπτονται από το υλικό που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και στην οδηγία για τη συγκριτική διαφήμιση θα πρέπει να βρούμε ποιες διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Εγώ επομένως σας σύστηνα τα θέματα αυτά να αντιμετωπιστούν μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας έκφρασης και όχι μέσα στα πλαίσια των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Um, θα ξανάρθω στο θέμα αυτό. Μικρόφωνο, μικρόφωνο παρακαλούμε. Αλλιώς δεν φαίνεστε στην εικόνα. Για να ξαναγυρίσω στον κανονισμό 2005-2006, τη συνεργασία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνε για την προστασία των καταναλωτών, βασίζεται στο ότι η συνεργασία δεν δίνει δικαιώματα στον ε, μεμονωμένο καταναλωτή, απλώς ρυθμίζει τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και βάσει έρευνα τη ευρωπαϊκή ε, επιτροπή λειτουργεί καλά, αλλά πολλές φορές είναι πολύ δάπανη αυτή η διαδικασία εφαρμογής σε διαμεθοριακό επίπεδο. Υπάρχει πάντα λοιπόν χώρος για βελτίωση και αν δεν λειτουργεί λοιπόν καλά η εφαρμογή, δεν φταίνε οι καταναλωτές, όπως φάνηκε στο παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Δεν είναι δεν βοηθάει πολύ τον καταναλωτή εάν δεν είναι καλή εφαρμογή. Και να έρθω στο επόμενο ερώτημα για το, τη μαύρη λίστα του παρατήματος 1 και την πλήρη εφαρμογή και το γιατί δεν δουλεύει καλά αυτή η μαύρη λίστα. Ο στόχος της είναι να δώσει κάποια, ε, κάποιες κατευθύνσεις στα εθνικά δικαστήρια για να ξέρουν ποια είναι, ποιες είναι αθέμητες πρακτικές και ποιες όχι. Αλλά και πάλι βέβαια δεν ευκολύνει πολύ τη θέση τους γιατί πρέπει πάντα να αποδείξουν ορισμένες από τις προϋποθέσεις του παραδείγματος 1 Παραδείγματος χάρη αναφερθήκατε στο θέμα της προστασίας των παιδιών που είναι πολλές φορές το αντικείμενο διαφήμισης που έχουν σε στόχο να υποχρεώσουν τους γονείς τους να αγοράσουν κάτι. Αλλά η οδηγία δεν αναφέρει ποιος είναι παιδί και ποιος δεν είναι, κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Υπάρχει επομένω κάποια ασάφεια <clears throat> και κάποια ανάγκη ερμηνείας στο σημείο αυτό. Επομένως αυτή η οδηγία σε αυτό το σημείο δεν ήταν τόσο επιτυχής όσο θα θέλαμε. Και για την πλήρη εναρμόνιση Η νομοθεσία στη Δανία είναι ίδια όπως και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Έχουν ήδη αποφασιστεί κάποιες, έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση δικαστική για κάποιες αποδείξεις. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές η πλήρης εναρμόνιση ξεπερνάει πολύ περισσότερο την εθνική νομοθεσία από ό,τι αναμενόταν καταρχήν και φαίνονται και περισσότερες ελλείψεις όπου τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν κάτι στην εφαρμογή της οδηγίας ή να βελτιώσουν την νομοθεσία τους και να την προσαρμόσουν στην οδηγία. Και ο συνάδελφός μου θα σας πει τα υπόλοιπα. Και ε, για το θέμα της ε, πρακτικής ε, των λεγόμενων City Guides είναι γνωστό σε εσά γιατί υπήρξε και εδώ μια έκθεση που μπορώ να σας υπενθυμίσω <clears throat> στην προηγούμενη οδηγία για τις ε, παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές διαφήμισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι οδηγοί, οι ίδιοι ορισμοί <clears throat> όπως και στην οδηγία για τις, για τις καταχρηστικές πρακτικές. Δηλαδή να αναφέρονται και σε σχέση μεταξύ επιχειρήσεων αυτές οι πρακτικές οι οποίες θεωρούνται μη θεμητές. Παραδείγματος χάρη αποστολή τιμολογίων που δεν είναι πραγματικά τιμολόγια, όπως ήταν η περίπτωση των City Guides. Γιατί με τον τρόπο αυτό πολλές μικρές εταιρείες τι χάνουν, γίνονται θύματα απάτης με αυτόν τον τρόπο. I think the two remaining questions relate. Τα δύο ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα έχουν να κάνουν με την προστασία των παιδιών και τους καταναλωτές στο eBay, πώς γίνεται διάκριση μεταξύ εμπόρων και επιχειρήσεων στο eBay και θα ήθελα να επανέλθω στο σημείο 28 του παρατήματος 1 που λέει ότι οποιαδήποτε διαφήμιση η οποία είναι παρότρινση προς τα παιδιά να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή να ταλαιπωρήσουν τους γονείς τους προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί αθέμητη πρακτική και υπάρχει και μια άλλη ρήτρα της οδηγίας για την προστασία των παιδιών και αυτό είναι το άρθρο 5, σημείο 2, β, που λέει ότι αν μια ειδική ομάδα καταναλωτών εμπλέκεται, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον είναι, έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, παραγωγός χάρη νέοι καταναλωτές, παιδιά, επομένω η οδηγία υποστηρίζει την ιδέα ότι μπορούν να υπάρχουν ειδικέ ομάδε καταναλωτών που απαιτούν ειδική προστασία, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί από τα δικαστήρια, δεν έχει ληφθεί υπόψη από τα δικαστήρια σε αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι μεταπολούν προϊόντα ή τα πουλούν στο eBay και σε αντίστοιχους οργανισμούς, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς πού σταματάει το καθεστώς ως καταναλωτή ενός πολιτή και πότε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια επιχείρηση. και το eBay είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτά τα προβλήματα του πώς καθορίζουμε ποιος είναι επιχείρηση και ποιος είναι καταναλωτής. Στη Γερμανία ο κανόνας είναι ότι οποιοδήποτε βγάζει ένα προϊόν στην, στο eBay θεωρείται ότι είναι <clears throat> μια επιχείρηση. Ήθελε κανείς άλλος να πάρει το λόγο, κάποιος από τους εμπειρογνώμονες ενδεχόμενα. Έχουμε και χρόνο στη διαθέσή μας, ε, αν ε, θέλετε να πείτε κάτι. Ο κύριος Απρομόντη ίσως ε, θα ήθελα να πάρει το λόγο. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θίξαμε τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και, την, και τον πυρήνα, αν θέλετε, των, των προβλημάτων εφαρμογής της οδηγίας. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, ακούστηκαν πολλά σχόλια, πρέπει να τα ε, εξετάσουμε να τα μελετήσουμε. Ούτως ή άλλως η εφαρμογή της οδηγίας στα θέμα των εμπειρικών πρακτικών αποτέλεσε και αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής μας σε μια άλλη θητεία. Ο κύριος Αβραμόντη θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας γιατί ζήτησε να συνταχθούν αυτές, τόσο, αυτές οι τόσο ε, σημαντικές και ενδιαφέρουσες εκθέσεις ε, για τις ε, εμπορικές πρακτικές online και για, και για το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας και επίσης οι εκθέσεις αυτές παρουσιάζουν και τις ε, ενδεχόμενες δυσκολίες και προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή. Πιστεύω ότι όλοι ευχαριστούμε τον κύριο Ζουβά για την, ε, για την έκθεσή του, για την ε, για τον αντίκτυπο της διαφήμισης της συμπεριφορά των καταναλωτών και πιστεύω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ε, συμμετέχουν και θα συνεργαστούν μαζί του. Τώρα, θα ήθελα να θίξω δύο συγκεκριμένα θέματα. Το ένα είναι το θέμα της νομικής ε, ε, σαφήνειας και ασφάλειας και το δεύτερο είναι το θέμα της εφαρμογής, της υποχρεωτικής εφαρμογής. Μία οδηγία εναρμονίζει πλήρως τις ουσιαστικές διατάξεις ενός κράτους μέλους που αφορούν τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές χωρίς να επιβάλλει αν θέλετε ένα σύστημα εφαρμογής στα κράτη-μέλη διότι οι νομικές πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ποικίλουν. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Γερμανία που αποτελούν την μειοψηφία, που έχει ένα καθαρά ιδιωτικό σύστημα εφαρμογής και μετά έχουμε άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία που έχουν ένα σύστημα κυρίως ε, δημόσιο εφαρμογής. Όπως ε, έχουμε πει και στην ανακοίνωσή μας σχετικά, ε, της προηγούμενης χρονιάς σχετικά με την εφαρμογή του, και κεκτημένου που αφορά τους καταναλωτές, η ουσιαστική εφαρμογή του ανταγωνιστικού δικαίου απαιτεί ένα σωστό μείγμα δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, όμως πάντα ο δημόσιος φορέας θα παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο. Πιστεύουμε ότι το ιδανικό θα ήταν οι μελέτες να λάμβαναν υπόψη και την εμπειρία κρατών που έχουν εφαρμόσει, που έχουν μεταθέσει έγκαιρα την οδηγία, όπως είναι η Ιρλανδία και η Ιταλία επίσης. Και οι δημόσιες αρχές εφαρμογής εκεί στις χώρες αυτή, αυτές έχουν εξασφαλίσει εξαιρετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες, προσπάθειές τους και έχουν ε, και συγκεκριμένα ε, πορίσματα, έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά για την νομική σαφήνεια και νομική ασφάλεια, μιλάμε για ένα οριζόντιο κείμενο, νομοθετικό κείμενο, το οποίο περιέχει και κάποιες ε, θεωρητικές έννοιες. Θεωρητικές έννοιες όπως ε, ε, η, εμπορική, η επαγγελματική επαγγελματική πείρα, η σαφήνεια κτλ. Υπάρχουν διάφορες έννοιες γενικότερα που χρειάζονται να αποσαφινιστούν. Πέρυσι η Κομισιό δημοσίευσε ένα κείμενο, το οποίο είναι ένα ζωντανό κείμενο, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς από την Κομισιό. Αναφέρομαι όμως και στην νομική βάση που προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρουσιάζουν, αν θέλετε, την νομοθεσία τους. Θα παρουσιάζεται η νομοθεσία των κρατών μελών και η νομολογία, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και όσο θα περνάει ο καιρός θα υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες υποθέσεις που θα υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλές υποθέσεις που ήδη έχουν, βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια νομική σαφήνεια ή ασφάλεια όσον αφορά το ε, περιεχόμενο της οδηγίας. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι λίγα κράτη-μέλη έχουν μεταθέσει έγκαιρα την οδηγία, τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, έχουν καθυστερήσει και κάποια κράτη έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Να ολοκληρώσω ε, μιλώντας λίγο για τη διασυνοριακή εφαρμογή υπάρχει ένας κανονισμός για την προστασία των καταναλωτών που δημιουργεί ένα δίκτυο φορέων που εφαρμόζουν την οδηγία, την νομοθεσία δηλαδή, και αυτοί ασχολούνται και με τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ούτως ή άλλως η οδηγία αναφέρεται στην προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος των καταναλωτών. Δεν μιλάμε για την διασφάλιση ε, του μεμονωμένου συμφέροντος ή του συμφέροντος του μεμονωμένου καταναλωτή. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε βέβαια και την ε, περισσότερο το διασυνοριακό χαρακτήρα της προστασίας του καταναλωτή, αλλά εάν οι αρχές... Μάλλον, εάν οι αρχές που ασχολούνται με την διασυνοριακή προστασία ενημερωθεί για την ε, αθέμητη αυτή πρακτική, τότε η αρχή αυτή θα μπορούσε να γίνει αίτηση βοήθειας στον αντίστοιχο φορέα, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο έμπορος. Επομένως, οι αρχές της χώρας προέλευσης, δηλαδή οι αρχές του κράτους του εμπόρου, θα πρέπει να ελέγξει τις πρακτικές και αν είναι αθέμητη πρακτική να τη σταματήσει. Όμως επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για την προστασία του συλλογικού συμφέροντος των, του καταναλωτή. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σας και τους ε, <clears throat> εμπειρογνώμονές μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή μας για να μπορέσει να αντλήσει κάποια συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να θέσει περαιτέρω ερωτήματα. Έχουμε χρόνο, αλλά ίσως είναι καλύτερα να <clears throat> επανέλθουμε ίσως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, αλλά σίγουρα θα ήταν χρήσιμο εισηγητή μα να αντλήσει κάποια συμπεράσματα και να μα αναφέρει το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στη σημερινή μα συνεδρίαση και στην προηγούμενη μα συνεδρίαση. Εγώ έχω αντλήσει μια σειρά από συμπεράσματα, τα εξή. Πρώτον, για τη σχέση μεταξύ διαφήμισης και κατανοητή υπάρχουν δύο σκόπελοι που πρέπει να τους αποφύγουμε. Καταρχήν το να δαιμονοποιούμε απόλυτα τη διαφήμιση. Είναι γνωστή αυτή η γελιογράφηση της διαφήμισης, αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Και ο δεύτερος σκόπελος, αν θέλετε, είναι μια αφελής προσέγγιση. Να, λέμε, να νομίζουμε ότι η διαφήμιση λέει πάντα την αλήθεια. Η διαφήμιση φυσικά είναι απαραίτητη είναι απαραίτητη ως ε, ένα είδος γράσου της οικονομίας, αυτό το οποίο βοηθάει την οικονομία να λειτουργεί και φυσικά προωθεί την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή με την προϋπόθεση ότι είναι θεμητή και ότι είναι διάφανη. Στην έκθεση πρωτοβουλίας μας, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, εμείς περιοριστήκαμε από το χρόνο και το χώρο ιδίως. Ο αριθμός των χαρακτήρων, όπως είναι γνωστό, είναι περιορισμένος. Επομένως, το να συντάξουμε μια έκθεση για τον αντίκτυπο στη διαφήμιση των καταναλωτή σε τρει ή τέσσερι σελίδε, μα υποχρεώνει να προβούμε σε επιλογέ. Οι επιλογέ αυτέ, κατά την άποψή μου, μπορούν να είναι εξή. Τονίστηκε πολλέ φορέ ότι υπάρχει το θέμα τη προστασία των πιο τροτών τμήματων του πληθυσμού. Και φυσικά ο νόμος σε όλες τις εκφάνσεις του έχει σαν στόχο να προστατεύσει κυρίως τους πιο ευάλωτους και εκεί πρέπει να αποδώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. <clears throat> Δεύτερον, και αυτό μου φαίνεται εξίσου και επίσης σημαντικό, οι τεχνικές και τα μέσα επικοινωνίας εξελίσσονται ραγδαία και η διαφήμιση επίσης εξελίσσεται ραγδαία. Ποιος θα πίστευε πριν από μερικές δεκαετίες ότι το να διαβάζει κανείς το προσωπικό σας ταχυδρομείο επιτρέπει σε ορισμένε εταιρείε να αντλούν τα συμπεράσματα για το πώς να έχουν καλύτερα στοχευμένη σε εσά διαφήμιση. Έχουν αναπτυχθεί επίσης τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία δημιουργούν μια μορφή διαφήμιση που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τις πιο παραδοσιακές εποχές διαφήμισης. Επομένως, η διαφήμιση στο διαδίκτυο θα είναι ο δεύτερος μεγάλος άξονας αυτής της έκθεσης σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της διαφήμισης στον καταναλωτή. <clears throat> Και τρίτον, πρέπει να υπάρχει και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Όσο εξευγενίζεται και γίνεται πιο λεπτολόγα η διαφήμιση και γίνεται πιο διεισδυτική, αλλά με τρόπο διακριτικό, κατά κάποιο τρόπο, τόσο περισσότερο πρέπει να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ο, <clears throat> ο καταναλωτής και να είναι ένας πολίτης ο οποίος θα είναι πεφωτισμένος σε σχέση με τα θέματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να υποστηρίξουμε μια ευρία ενία παιδαγωγική προσέγγιση προς τον καταναλωτή. Όλα αυτά τα γνωρίζει η Κομισιόν πιστεύω. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν όταν γίνει η αξιολόγηση της ε, οδηγίας αυτής για τις ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές, θα πρέπει να αντιλήσει τα κατάλληλα συμπεράσματα η Κομισιόν και αυτό είναι και ο δικός μας στόχος, <clears throat> εν μέρη χάρη στο έργο σας, ε, μέλη, του πάνελ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται η πρώτη παρουσίαση της έκθεσής μου στην Επιτροπή μας στις 13 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Η καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες αρχές Οκτωβρίου 5 Οκτωβρίου νομίζω έχει προταθεί σε αυτήν την περίπτωση και θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή μας <clears throat> στις 26 ή 27 Οκτωβρίου, δεν ξέρω αν αυτό σας βρίσκει σύμφωνο κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να προσαρμοστούν στη βάση της ορίμανσης των απόψεων στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Προσβλέπουμε σε αυτές τις επόμενες φάσεις θα προσπαθήσουμε με το χρονοδιάγραμμα να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσουμε το περιεχόμενο αυτής της σημαντικής έκθεσης. Ενδιαμέσως οι μελέτες αυτές και έχω πάρα πολύ υλικό εδώ πέρα το οποίο θα σας βοηθήσει και σε θέματα εναρμόνισης και της έκθεσης για τα θέματα των καταναλωτών που εκπονεί ο κύριος Σφάμπ. Ήταν πολύ χρήσιμο το ότι ο κύριος Αβρομόντε μας υπενθύμησε ότι του χρόνου η Κομισιόν θα κάνει μια επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας για, την, ε, για τις αθέμητες πρακτικές. Είναι κάτι που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας και κάποιοι συντονιστές ίσως θα θέλουν να το γράψουν στην ατζέντα τους για του χρόνου. Επομένως, αυτό το έγγραφο θα είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα άτομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες μας και πάλι για τη συμβολή τους σε αυτή τη διαδικασία και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξανακαλέσουμε να συμβάλλουν στο έργο μας που αφορά την προστασία των καταναλωτών και το οποίο θα εκτυλιχθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών περίπου. Μπορώ λοιπόν να κλείσω αυτή τη συνεδρίαση. Η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει στις 3 ώρα το απόγευμα σας υπενθυμίζω ότι είμαστε σε μια άλλη αίθουσα. Είμαστε στην Α3Ε2 στο κτίριο Αλτιέρο Σπινέλη. Θα σας παρακαλέσω να πάρετε λοιπόν όλα τα έγγραφά σας. Έχουμε δύο θέματα. Στις τρεις συζητούμε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για την τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά στις 4 παρατέτατο ο, και, ο κύριος Παντσέρη θα παρουσιάσει την ε, το θέμα του εμπορικού δικαίου και οικογενειακού δικαίου στο πρόγραμμα της Στοκόλμης. Ελπίζουμε να τελειώσουμε 4.30. Γεια σας.